We maintain the vote open because our colleagues are... Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία, διότι έρχονται ακόμα συνάδελφοι. Everybody have voted. Ψηφίσατε όλοι. Κύριε Σκερβάντη. Ωραία. Όχι. Έχουμε μία ψήφο παραπάνω από τους φιλελεύθερους. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Adesso votiamo. Ε, και τώρα ψηφίζουμε την συμβιβαστική που έχει επιτευχθεί με το Συμβούλιο για την ε, πρόταση οδηγίας ΝΕΚ η είναι η συνάδελφος Γκέρλινγκ. Για αυτή τη συμφωνία λοιπόν ψηφίζουμε. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ένσταση στο, με βάση το άρθρο 106 για την παράταση της περίοδου χρήσης ε, αδειοδότησης μάλλον της γλυφοσάτης το επέβαλε η συνάδελφος Κιλόνεν. Άρχισε η ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία μάλλον. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα και περνάμε στην προφορική ερώτηση για τα τρανς λιπαρά. Προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ψηφίζουμε τώρα την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Πάντοτε για τα ε, τρανσλιπαρά άρχεται. Ψηφίζετε όλοι. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ερώτηση για την COP22 Μαρακές. Αλλά πρώτα-πρώτα ερώτηση προς την Κομισιόν. Άρχεται. Πέρας. Γίνεται. Τώρα, ερώτηση προς το Συμβούλιο. Άρχεται. <coughs> Avete votato tutti, il voto è... Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται. Food Contact Material. Σάλτερ Μόζε είναι η συγγήτρια. Η αρμόδια του επιτροπή είναι δική μας. Και ξεκινάμε με την ε, τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 42 υπέρ κατά απόχέ συγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 7 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασ... Ε, τροπολογία, με συγχωρείτε, 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, όχι. Ε, εντάξει, πάντως συγκρίνεται ούτε ή άλλως. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 83 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός. Avete Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 84. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Συγκρίνεται. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την 94. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Αποχές έλεγχος. στι ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 96. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3α συμβιβαστική, 3α υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, ε, συγγνώμη, τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 116. Ως link. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 121. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 120 υπέρ. Α, καταπίπτει. Τι πρέπει να ψηφίσουμε την 116, ε, 117 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τώρα ψηφίζουμε την ε, συμβιβαστική 3β υπέρ αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 29 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται τώρα ψηφίζουμε την ε, τροπολογία 132. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 134. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της πληροφορια Απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές έκρινεται 138 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίσατε όλοι Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το 139 πιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 9 υπέρ, κα, υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Τροπολογία 158 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τις... τα εκτιμώντας. Τροπολογία 11 για τα εκτιμώντας α. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 18, ποιοτικά είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκαίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία τώρα 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34. 34 έχει καταπέσει. Την 35 πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Έκρινεται. Ψηφίζουμε την 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία ε, άρχεται. Avete Ψηφίσατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 17 της ημερησίας μας διάταξης που είναι η ψηφοφορία για την ε, ασφάλεια για τις ε, εξορίξεις ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανοιχτή θάλασσα, τροπολογία 1 υπερκατά, αποχές, έλεγχος. Avete votato tutti? Ψηφίζετε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο 5 Έχουμε προφορική τροπολογία της συναδέλφου Ριβαζή. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε με την ε, προφορική. Την τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. No, I gruppi non erano nemmeno convinti. Quindi avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τριχοσυμφιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε την 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 ε, υπέρ κατά αποχές ε, έλεγχος. Ψηφίζατε όλοι. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σε τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές Ε, 5. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές οι σοσιαλιστές δεν κατάλαβα να είστε υπέρ μάστε εγκρίνεται έλεγχος άρχεται απορρίπτεται ε, συμβαστική 10 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση τροποποιημένη. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το σημείο 18 της ημερησίας διατάξεως. Στόχοι κλειδιά για την 16η ε, Σύνοδο των Μερών ΣΥΤΕΣ. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Avete Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Αγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Respinto. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές έγκαινεται έλεγχος Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Ναι. Τέλο ε. ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 έχει καταπέσει και πάμε στην τροπολογία 32. Και αυτή έχει καταπέσει ή όχι. 31. Και η 32 λοιπόν έχει καταπέσει. Πάμε στην 33 υπέρ. Κατά αποχές ε, Για την τροπολογία 34 έχουμε μία προφορική του ΕΛΚΑ που σας τη διαβάζω υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Κομισιόν και των κρατών μελών να συμφωνήσουν για ε, παγκόσμιες κατευθύνες γραμμές όσον αφορά την την, ε, το trophy hunting έτσι ώστε να μην ε, ε, για να προστατευτούν εκείνα τα είδη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα 2. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Μα ψηφίζουμε λοιπόν με την προφορική του ΕΛΚΑ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη 35. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ναι, 38. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 40. 40 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά <coughs> αποχές έλεγχος. Avete votato tutti, voto è chiuso. Ψήφισατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα η τροπολογία 50. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 53 δεν την ψηφίζουμε. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά έλεγχος Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 32-32. Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα ψηφίζουμε για την 76 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε unblock τη 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 και 89. Υπέρ. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε στην τροπολογία 90 έχουμε προφορική του ΕΛΚΑ. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική αυτή η τροπολογία. Όχι. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 90 όπως τροποποιείται με την προφορική υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την αρχική εκδοχή του 90 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ε, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, unblock τις τροπολογίες 91 μέχρι και 90, 92 και 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Έλεγχος. Votiamo adesso. Ah, eh, ok. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε προφορική του συναδέλφου Αφρόντε. Θέλω να μας εξηγήσετε το περιεχόμενό της. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό ε, το είδος είναι ένα μικρό ψάρι που ζει σε πολύ περιορισμένη περιοχή. Της δεκαετία του 90 ανακαλύφθηκε ως είδος για τα ενιδρία ο πληθυσμό μειώθηκε κατά 20% και τα τελευταία χρόνια 40% μειώθηκε ε, η πίβερξή του. Ήδη είναι σε είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση και γι' αυτό θέλουμε να μετακινηθεί από το παράρτημα 2 του ΣΥΤΕΣ στο 1 που το προστατεύει πιο αποτελεσματικά. Δεν αναπαράγεται δε σε συνθήκες ενιδρίου. Μάλιστα. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίζουμε την ε, προφορική λοιπόν υπέρ, κατά, αποχέσει, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας της ε, ψηφοφορίας, εγκρίνεται ε, τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 α όχι συγγνώμη καταπίπτει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 Uh, Έχουμε μια σύντομη διακοπή της συνέδριασή μας. Ξεκινάμε... Uh, minutes before 11. παρα 2 λεπτά, γιατί έρχεται ο Υπουργό Υγεία τη Σλοβακική Προεδρία που έρχεται να μα παρουσιάσει τι προτεραιότητε εδώ στην Επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασής μας. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τόμας Ντρούκερ, Υπουργό Υγείας της Σλοβακίας, που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Προεδρίας του Συμβουλίου. Καλωσορίζουμε την νέα Προεδρία του Συμβουλίου και δίνω το λόγιο στον κύριο Τόμας Τρούκερ για να μας ε, κάνει την εισαγωγική του ομιλία και κατόπιν θα προχωρήσουμε στη συζήτηση. Συνήθως έχουμε δύο γύρους ερωτήσεων, ε, τον πρώτο με ε, τους ε, εκπροσώπους των ε, πολιτικών ομάδων και μετά δίνουμε τον λόγο και στους ε, υπόλοιπους ευρωβουλευτές και θα έχετε την δυνατότητα να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΕΝΒΗ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής αυτής. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Σλοβακικής Προεδρίας στον τομέα της υγείας. Το 2016 είναι η 12η επέτειος της ε, προσχώρησης της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η πρώτη φορά που η Σλοβακία θα κατέχει ηγετικό ρόλο στο Συμβούλιο. Έχουμε αναλάβει την Προεδρία σε δύσκολη εποχή όπου αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις όλοι μας. Μπορεί να προκύψουν αναπάντεχα ζητήματα και μάλιστα αυτό συμβαίνει πιο συχνά τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Ό,τι και να γίνει όμως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Παρά τις προκλήσεις αυτές, και την ε, αυξανόμενη αβεβαιότητα, η Προεδρία της Σλοβακίας ε, σκοπεύει να προωθήσει ένα θετικό θεματολόγιο και να ενισχύσει τις ε, βιώσιμες λύσεις. Οι στόχοι της Προεδρίας μας μπορούν να επιτευθούν με στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατηρήσουμε το θετικό και δυναμικό πνεύμα κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργαστούν πάνω σε σημαντικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθά τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσφέρει πρακτικές λύσεις στις καθημερινές ζωές τους. Σημαντικό όμως είναι επίσης ότι πρέπει οι άνθρωποι να, να καταλαβαίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ε, τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ήταν η κινητήρια δύναμη για την πρόοδο και πάντα έχει υπερασπιστεί τα ε, συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη και η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την μελλοντική διαμόρφωση της πολιτικής υγείας είναι ζωτικής σημασίας είσαστε οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος σας ως συνομοθέτες είναι αποφασιστικός ε, για την υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Πρωτού σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Προεδρία των Κάτω Χωρών για την σκληρή δουλειά τους ε, και την βοήθεια τους ως εταίροι μας στο τρίο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βασιστούμε στα δικά τους επιτεύγματα και να πετύχουμε ε, να υπάρχει συνέχεια όσον αφορά το θεματολόγιο μας. Ε, στον ε, νομοθετικό τομέα η Σλοβακική Προεδρία μετά από τέσσερα χρόνια σκληρή δουλειά πάνω στα γιατροτεχνολογικά βοηθήματα και τα in vitro διαγνωστικά γιατρικά βοηθήματα σημειώνουμε με προεδρία ότι έχει επιτευχθεί, ε, σημειώνουμε με ε, ικανοποίηση ότι έχει επιτευχθεί η συμφωνία στις 15 Ιουνίου. Η Σλοβακική Προεδρία θα πρέπει να ε, κυρώσει τη συμφωνία αυτή στο Συμβούλιο και σκοπεύουμε να υποβάλουμε και τα δύο κείμενα στο Συμβούλιο για να υπάρξει πολιτική συμφωνία το Σεπτέμβριο. Χάρη στα επιτεύγματα της Ολλανδικής Προεδρίας έχουμε ε, ένα θέμα που, στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια στον τομέα της υγείας και είναι ο κανονισμός 726 του 2004. Ε, αποτελεί μέρος του πακέτου κτηνιατρικών μέτρων και θα προσαρμόσουμε την ταχύτητα πάνω στο θέμα αυτό στην πρόοδο στα άλλα κτηνιατρικά ε, θέματα. Επίσης, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή ανάμεσα σε αυτόν τον κανονισμό και το πακέτο νομοθετικών μέτρων στον κτηνιατρικό τομέα για να βρούμε τα ε, κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των μέτρων που θα πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με τον κανονισμό 726-2004. Όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα και την ασφάλεια των τροφίμων, Μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε όλη η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η νομοθεσία που εκπονείται αυτή τη στιγμή, να εφαρμόζει μια ενιαία προσέγγιση ε, από τη γεωργική εκμετάλλευση στο τραπέζι του καταναλωτή. Ήδη, υπά... Ήδη έχουμε αναφέρει ένα σημαντικό πακέτο, μια σημαντική δεσμή μέτρων στον τομέα αυτών την πρόταση για τα ακτινιατρικά φάρμακα και την πρόταση για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Ενώ η πρόταση για τις φαρμακούχες ζωοτροφές καλύπτεται από την Επιτροπή Άγκρη, αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Άγκρη, η πρόταση για τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι πολύ σημαντική για τη δική σας Επιτροπή. Να σας ενημερώσω ότι η Προεδρία της Σλοβακίας θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω ε, στο θέμα αυτό στα, στους προπαρασκευαστικούς σχηματισμούς του Συμβουλίου ο, με στόχο μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας να έχουμε μία εντολή που να αποτελέσει βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο και αποφασιστική σημασία ε, όχι μόνο για τον κτηνιατρικό, τον γεωργικό ε, τομέα και για τα κατοικίδια ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την δημόσια υγεία σε ε, της σχέσης του θέματος αυτού με την ε, μικροβιακή αντοχή που αποτελεί σημαντική πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά το θεματολόγιο υγεία, σε μια άλλη από τι προτεραιότητε ε, τη Σλοβακική Προεδρία στον τομέα εκτό τη νομοθεσία θα είναι η διαθεσιμότητα και η ελλείψει φαρμάκων. Κάτι που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για του ασθενεί στην Ευρώπη. Έχουν ε, ακουστεί φωνές που μιλούν για έλλειψη φαρμάκων ε, σε διάφορα κράτη-μέλη. Ε, έχουν ακουστεί αυτά και από πλευράς ενώσεων ασθενών καθώς και από επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Για μένα είναι σοβαρό το θέμα αυτό και στόχος είναι να υπάρχει επαρκές επίπεδο ιατρικής περίθαλψης καθώς και πρόσβαση στα φάρμακα για τους ασθενείς. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα φάρμακα δεν είναι κανονικά αγαθά όπως όλα τα άλλα, λόγω της σημασίας τους για τη δημοσία υγεία και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση στα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, ελλείψεις, ε, άσχετα από αν αυτές οφείλονται σε στην, με, με, στην παραγωγή ή στις ε, εξαγωγές. Στην ε, ομάδα εργασίας για τη δημόσια υγεία σε ανώτερο επίπεδο καθώς ε, και στις, στην άτυπη υπουργική συνεδρίαση στην Πρατισλάβα θα προωθήσουμε τη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Επίσης, αναγνωρίζουμε τη σημασία της πολιτικής κατά του καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, που βρίσκεται επικεφαλής στην ε, παγκόσμια συζήτηση για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού. Η Προεδρία της ε, Σλοβακίας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε και κατά την 7η διάσκεψη των μερών της Σύμβασης Πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού στην Ινδία φέτος να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουμε συντονισμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα θέματα του θεματολογίου της συνάντησης αυτής. Συνεχίζω όσον αφορά τι προτεραιότητέ μα. Το Συμβούλιο, όπω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρεί το πρόβλημα τη μικροβιακή αντοχή σοβαρό και έχει καλέσει τα κράτη-μέλη επανειλημμένα να εργαστούν σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Η Προεδρία της Σλοβακίας θέλει να ασχοληθεί με το θέμα της φυματίωσης και της ανθεκτικής σε πολλά φάρμακα φυματίωσης. Η φυματίωση και τα πολυανθεκτικά βακτηριακά στελέχη της φυματίωσης ε, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την υγεία και η φυματίωση συνδέεται επίσης με συνοσυρότητες ε, σε σχέση με άλλες ασθένειες ε, όπως είναι το ε, AIDS. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ομάδας εργασίας για τη δημόσια υγεία σε ανώτερο επίπεδο στις 15 Ιουλίου του 2016 η Σλοβακική Προεδρία θέλει να ξεκινήσει την συζήτηση για να υπάρξει ένα πιθανό πλαίσιο πολιτικής για την φυματίωση, το AIDS και την ε, υπατήτηδα σε. Κατόπιν θα ακολουθήσει η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Υγείας στην Πρατισλάβα στις 3 και 4 Οκτωβρίου του 2016. Οι μεταδοτικές ασθένειες έχουν επηρεαστεί από δύο σημαντικές γιατρικές εφευρέσεις, ε, ε, τον εμβολιασμό και τα αντιβιωτικά. Τα εμβόλια βρίσκονται μπροστά από τα αντιβιωτικά κατά κάποιο τρόπο, διότι τα αντιβιωτικά ε, χρησιμοποιούνται ε, μετά την εμφάνιση μιας νόσου, ενώ ο εμβολιασμός ε, προλαμβάνει την εμφάνιση της νόσου. Και τα αντιβιωτικά σκοτώνουν τα μικρόβια, ενώ τα εμβόλια έχουν στόχο τους ιούς. Η Προεδρία θεωρεί ότι το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού είναι σημαντικό εργαλείο στην ε, καταπολέμηση της υπερβολικής κατανάλωσης αντιβιωτικών και γι' αυτό θέλει να ε, ευαισθητοποιήσει τον κόσμο ε, για, τον εμβολιασμό. Πόσο μάλλον που υπάρχει αυξανόμενη τάση εκστρατιών κατά του εμβολιασμού. Η Σλοβακική Προεδρία θα ασχοληθεί με το θέμα του εμβολιασμού κατά την ε, άτυπη συνάντηση Υπουργών Υγεία ε, στην Πρατισλάβα. Άλλο θέμα που προκαλεί ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, το υπερβολικό βάρος, κάτι που έχει η παχυσαρκία που έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ το 1995 υπήρχαν 200 εκατομμύρια ανθρώπων υπέρβαρων ή παχύσαρκων σε όλο τον κόσμο, ε, σήμερα ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια, το 2000 μάλλον. Ε, το υπερβολικό βάρος, ε, η υπερβολική πρόσληψη θερμίδων, τα χωρισμένα λιπαρά, τα τρανς λιπαρά, η ζάχαρη και το αλάτι, καθώς και η χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και προϊόντων ολικής αλέσεως έχουν οδηγήσει σε κακή και σε συνήθειες. Και πιστεύουμε ότι ο επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης των τροφών ε, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ε, για να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου, όπως είναι τα κορεσμένα λιπαρά, τα τρανς ε, λιπαρά, η ζάχαρη και το αλάτι. Και γι' αυτό η Σλοβακική Προεδρία θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη-μέλη και θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην καλύτερη διατροφή και την μείωση της εμφάνισης των μη μεταδοτικών ασθενειών. Οι μη μεταδοτικές ασθένειες αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ασθενειών στην Ευρώπη και είναι υπεύθυνε για το 86% όλων των θανάτων. Επηρεάζουν πάνω από το 80% των ε, ανθρώπων άνω των 65 ετών και αποτελούν σημαντική πρόκληση για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών. Οι καλές ε, συνήθειες ε, ο υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να μειώσει την ε, ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και έτσι να μειώσει το κόστος ε, της ε, περίθαλψης και να οδηγήσει σε περισσότερη ανάπτυξη και παραγωγικότητα. Φιλοδοξία της Προεδρίας μας είναι να ενισχύσουμε τους στόχους και τις δραστηριότητες στον τομέα των χρονίων μη μεταδοτικών ασθενειών και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης των τροφών και την μείωση των παραγόντων κινδύνου. Για να το πετύχουμε αυτό, η Προεδρία μας ε, θα οργανώσει μία διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την ε, πρόληψη όσον αφορά τις μη μεταδοτικές ασθένειες ε, και την ε, πρόθεση ε, της, του υγιεινού τρόπου ζωής στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου του 2016 στην Πρατισλάβα για να συζητήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την μείωση των παραγόντων κινδύνου και την καλύτερη διατροφή. Πολλές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν θέσει την άνοια ως προτεραιότητα και έχουν ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι το, μέχρι το 35% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρει από διαταραχές ε, του εγκεφάλου. Και το κόστος ε, από τις ε, παθήσεις αυτές αντιπροσωπεύει το 24% των συνολικών δαπανών για την υγεία στην Ευρώπη το 2010. Στην Ευρώπη το κόστος ε, των ε, παθήσεων αυτών είναι υψηλότερο από ότι για άλλες ασθένειες όπως είναι οι ε, καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. Το έμεσο κόστος είναι επίσης πολύ σημαντικό και είναι πολύ πιο δύσκολο να υπολογιστεί. Ε, και συμπεριλαμβάνει την ε, μείωση της ε, παραγωγικότητας, την αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, καθώς και των συγγενών του, καθώς και το κοινωνικό στίγμα με το οποίο συνδέεται. Για την προτεραιότητα αυτή η Προεδρία μας οργανώνει μια διάσκεψη στις 29 Νοεμβρίου στην Πρατισλάβα ε, πάνω στην νόσο του Αλσχάιμερ για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτών ε, για να ασχοληθούμε με τις επιστημονικές, ιατρικές και κοινωνικές στοιχείες ε, της άνοιας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Επικροτώ την δυνατότητα που μου δόθηκε σήμερα να σα ενημερώσω σχετικά με τις προτεραιότητε της Προεδρίας τη Σλοβακία στον τομέα τη Υγεία και να απαντήσω σε ερωτήσει. Σα Ευχαριστώ. you. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Να αρχίσουμε με τον πρώτο γύρο των τοποθετήσεων με τους συντονιστές δηλαδή. Πέτερ Λίζε για λογαριασμό του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσά κύριε Προεδρεύον για την ανάπτυξη της, ε, του θεματολογίου σας. Μιλήσατε για τις αντοχές σε αντιβιωτικά. Είναι προτεραιότητα για μας. Έχουμε και την νομοθετική διαδικασία την οποία παρακολουθεί ως εισηγήτρια η Φανσουάζ Γκροστέτ της πολιτικής μας ομάδος. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα που απασχολούν ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο. Αφενός, <coughs> Η μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών. Στην έκθεση που απαντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνεται μάλλον, ή μάλλον στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνεται μόνο η στην προταση της ευρωπαικης επιτροπης περιλαμβανεται μονο η καταγραφη των αντιβιωτικών που χορηγούνται στον γεωργικό τομέα. Και από την καταγραφή αυτή θα πρέπει να συναχθούν κάποια συμπεράσματα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να υποστηρίξετε τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Δεύτερο και πιο γενικά, για τις αντοχές σε αντιβιωτικά στην ιατρική ανθρώπων να βάλετε κάποιες προτεραιότητες για τις ε, μη μεταδοτικές ασθένειες, για όλους μας ασφαλώς αποτελεί προτεραιότητα. Από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος νομίζω δεν πρέπει να επισέλθουμε σε υπερβολική λεπτομέρεια στις νομοθεσίες που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους να αποκομίσουν την εντύπωση ότι τους υπαγορεύουμε τι θα καταναλώνουν, τι θα τρώνε και τι όχι. Μιλούμε περισσότερο για την διατροφική αξία. Η Επιτροπή μας προημερών αλλά και οι ε, Ολομέλη απέριψαν αυτά τα διατροφικά προφίλ. Νομίζω ότι και εσείς θα πρέπει να σεβαστείτε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή να χορηγηθούν με πληροφορίες στους ε, πολίτες, όχι όμως να τους υπαγορεύσουμε τι θα τρώνε και τι δεν θα πρέπει να τρώνε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των σοσιαλιστών. Κύριο Πανιού, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση και την σύνοψη των προτεραιοτήτων που επιθυμείτε να χειριστείτε σε θέματα υγείας υπό Σλοβακική Προεδρία. Τρία θέματα. Πρώτο, η ε, νομοθεσία σχετικά με τη ρύθμιση των καινοτόμων φαρμάκων, για τις τιμές δηλαδή των καινοτόμων φαρμάκων. Στο πρόγραμμά σας, αλλά και ε, ακολουθείτε τις γραμμές της Ολλανδικής Προεδρίας για την πρόσβαση στα φάρμακα και ιδίω για την ρύθμιση των τιμών των καινοτόμων φαρμάκων. Θα πρέπει να εγκρίνουμε σύντομα διεθνή νομοθεσία που να φροντίζει, να γίνει αντιληπτό δηλαδή, ότι τα καινοτόμα φάρμακα δεν είναι απλά καταναλωτικά αγαθά και ότι χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στους αρρώστους. Και ε, θα επαναφέρεται την συζήτηση για τη νέα οδηγία για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποσύρει την νομοθετική της πρόταση τον Δεκέμβριο του 2014, διότι δεν προβλεπόταν συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Ευρωπαϊκή νομοθεσία όμως σε αυτό το ε, τομέα προτεραιότητας μας φαίνεται αναγκαία. Δεύτερο, η αναγκαστική, η δεσμευτική ε, αναφορά της προελεύσεως του κρέατος στα ε, προπαρασκευασμένα τρόφιμα. Όσο γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ μιας υποχρεωτικής ιχνηλασιμότητας του κρέατος και του γάλακτος που περιλαμβάνεται σε ε, προπαρασκευασμένα τρόφιμα. Είναι προτεραιότητα αυτή για τον φάκελο υγεία της, προεδρία της Προεδρίας σας. Και εάν ναι, θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα επιβάλλει τη συστηματική αναφορά της προελεύσεως γάλακτος και κρέατος. Τρίτο, ο καπνός. Στο πρόγραμμά σας λέτε ότι θα αποδώσετε την αναγκαία προσοχή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την τρίτη διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον καπνό που θα γίνει τον Νοέμβριο του 2016 στην Ινδία. Έχει μεν κυρώσει το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 26 ε, Ιουνίου μάλλον του 2016 και έτσι φτάνουν τα 19 μέλη που έχουν κυρώσει. Τι θα γίνει με τις χώρες μέλη που ακόμα δεν έχουν κυρώσει για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να έχει ε, κυρωθεί από 40 συμβαλόμενα μέρη. Και υπάρχει και μεγάλη ανισότητα σε ζητήματα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον καπνό. Χώρες όπως Αυστρία, Φιλανδία, Γαλλία έχουν τονίσει ότι υπάρχει αναγκαιότητα να προκληθεί μεγαλύτερη σύγκληση των φορολογικών συντελεστών κατανάλωσης ε, για τα προϊόντα καπνού θα υποστηρίξετε τις χώρες αυτές στην θέλησή τους να καταλήξουν σε μεγαλύτερη σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των τιμών του καπνού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και αναμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευρωπαίοι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ, η ε, Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ερωτώ για την στάση σας για το γενικότερο policy making και τι αξία θα δώσετε στις επιστημονικές συμβουλές. Έχουμε διεξαγάγει πολλές συζητήσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και ιδίως για τις χημικές ουσίες, αλλά όχι μόνο. Χθε διεξήχθη συζήτηση και όχι για πρώτη φορά αλλά ούτε και για τελευταία και ένα από τα θέματα που έχουν πολύ έντονη σχέση με την υγεία και ιδίω με οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι συνδεόμενοι οργανισμοί, είναι εάν θα χορηγήσουν συμβουλές προς εμάς, τους νομοθέτες, ή πάντως θα μας παράσχουν συμβουλές, που ενδεχομένως θα είναι, ε, δεν θα ε, συντεριάζουν με άλλες επιστημονικές συμβουλές και στο επίπεδο των χώρων μελών αλλά και στο ενωσιακό επίπεδο. Έχετε την πρόθεση στη διάρκεια της Προεδρίας σας να επιληθεί του θέματος αυτού και ενδεχομένως να το προωθήσετε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις στο πολιτικό επίπεδο βασισμένοι σε στέρεες επιστημονικές συμβουλές. Διότι νομίζω ότι αυτό, αν επιτύχει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Ευχαριστώ ε, κυρία συνάδελφε, η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Και εκ μέρου λοιπόν των φιλελευθέρων σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία σας και αναμένω με ενδιαφέρον την συνεργασία μαζί σας. Αναφέρατε διάφορα σημαντικά πράγματα που θέλετε να χειριστείτε στην διάρκεια της Προεδρίας σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα προσπαθήσουμε ασφαλώς να σας υποστηρίξουμε λόγω της σημασίας των θεμάτων αυτών. Σύντομη παρατήρηση για τις ιατρικές συσκευές. Είπατε ότι οι Σλοβάκοι θα προσπαθήσουν να δώσουν επίσημη μορφή στη συμφωνία στο Συμβουλίο. Μετά από μακρά διαδικασία βεβαίω. Δυστυχώ οι Ολλανδοί δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το θέμα, διότι υπήρχε ακόμα ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα είστε λοιπόν εσεί σε θέση να το ολοκληρώσετε. Είναι πάντως σημαντικό για όλου του ασθενεί στην Ευρώπη να έχουν δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια στο θέμα αυτό. Άλλο θέμα, μιλήσατε για τα κτηνιατρικά φάρμακα νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Στα πλαίσια δε αυτά μιλήσατε και για την αντοχή στα αντιβιωτικά. Έχω ένα θέμα εδώ. Μιλήσατε για την αντοχή στα αντιβιωτικά, των βακτηρίων δηλαδή, που θέλετε να προωθήσετε. Η Ολλανδή Υπουργό Υγεία τόνισε ιδιαίτερα το θέμα αυτό και έχει κάνει και πολλέ εκστρατείε διαφωτίσεως. Εσείς λέτε ότι θέλετε να το συνεχίσετε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά και εθνικέ στρατηγικέ, όπω έχουμε μία στη Γερμανία, θέλετε και αυτέ να τι συμπεριλάβετε. Όμω, στην ημερήσια διαταξή σα, στο θεματολογιό σα δηλαδή, έχετε και άλλα χρήσιμα πράγματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορούν αυτά να συνδυαστούν. Μιλήσατε για παράδειγμα για την οροθετικότητα, μιλήσατε για τη φυματίωση και ούτω καθεξής. Αυτή η διάσκεψη του Οκτωβρίου αναφέρεται μονάχα στις δύο αυτές ασθένειες ή και στην αντοχή των βακτηρίων στην, στα αντιβιωτικά. Νομίζω αυτό πρέπει να συνεχιστεί, διότι ανοίγουν και νέα πράγματα στην έρευνα. Για παράδειγμα, στην έρευνα στα ζώα. Χρησιμοποίηση, για παράδειγμα, καλών βακτηρίων κατά κακών βακτηρίων σε ορισμένες ζωονόσους. Συμπληρωματικά διατροφής των ζώων, τα οποία καθιστούν μετά περιττή την χρήση αντιβιωτικών. Αυτά όλα πρέπει να συνυπολογιστούν στη στρατηγική αυτή. Γι' αυτό, αυτό το νόημα έχει η ερώτησή μου, πόση σημασία αποδίδεται στα θέματα αυτά. Τώρα, για την παχυσαρκία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ χρήσιμο να προβούμε σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Όμως ταυτόχρονα να υπάρχουν και έγκαιρες πληροφορίες για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Για παράδειγμα, πρέπει να χορηγούνται συμβουλές ήδη στην περίοδο της κοίησεως, αλλά ακόμη και στα παιδιά των υπηαγωγείων. Μία εξειδικευμένη ερώτηση τώρα για ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρατε. Σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουμε για τον υδράργυρο και μία στρατηγική για την χρήση του ή μη χρήση του. Ποια είναι λοιπόν η θέση σας απέναντι στην ομοιοπαθητική ή εναλλακτική ιατρική όπου ο υδράργυρος σε μικρές βέβαια ποσότητες είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται. Το ίδιο στην ανθρωποσοφική ιατρική και γι' αυτό είναι χρήσιμο αυτές οι ιατρικές να έχουν πρόσβαση στον υδράγυρο. Ποια είναι η θέση σας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας σας. Έχουμε ακούσει ήδη πολλά για αυτές και πιστεύω ότι θέματα όπως η αντοχή στα αντιβιωτικά και άλλα θα συνεχίσετε να τα χειρίζεστε με τον τρόπο που έχουν ήδη αρχίσει οι προηγούμενες προεδρίες και σε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπατε σωστά, ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει η προτεραιότητά σας, διότι είναι κατεπήγον θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω όμως και ένα άλλο θέμα, το οποίο μου φαίνεται ακόμα πιο κατεπήγον δηλαδή τη ε, διαθεσιμότητα φαρμάκων στην αγορά. Το πρόβλημα δεν σημειώνεται μόνο στη Σλοβακία αλλά και στην Τσεχική Δημοκρατία και είναι μάλιστα τόσο σημαντικό που ε, άνθρωποι με ογκολογικά προβλήματα δεν έχουν έγκαιρη πρόσβαση στα φάρμακα. Δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία εν τέλει δεν είναι τόσο ε, δαπανηρά αλλά δεν είναι γενώσιμα. Παρόλο που εισάγονται τα πρωτότυπα φάρμακα στην Τσεχική Δημοκρατία αμέσως επανεξάγονται σε δυτικέ χώρες από τις τσεχικές αρχές, όπου είναι πολύ πιο ακριβά. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται εδώ για μια ικτρή αποτυχία της αγοράς. Πρόκειται για ένα αυξανόμενο πρόβλημα που έχει προκαλώσει τρομερή αναστάτωση στις χώρες μας και βασίζεται βεβαίως ε, στην θέσπιση τιμών των φαρμάκων, στο πρόβλημα δηλαδή αυτό που προκαλείται από τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων. έχετε περιλάβει τη δυνατότητα επανεξαγωγή στην νομοθεσία μας, χωρίς να υπάρχουν ποσοστά των φαρμάκων που μπορούν να επανεξάγονται. Όχι μόνο λοιπόν να μιλήσετε για το θέμα αυτό, αλλά να προτείνετε ειδικά μέτρα στι χωρέ μέλη. Διότι το πρόβλημα γίνεται χειρότερο με κάθε χρόνο που περνάει. Και τελικώς η συνέπεια είναι ότι οι ασθενείς δεν έχουν στη διάθεσή τους τα φάρμακα που χρειάζονται για την περίπτωσή τους. Αυτό λοιπόν όπως είπα είναι μοιραίο για ολόκληρο το σύστημα υγείας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα σημαντικά προβλήματα. Όμως νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σοβαρό. Δεν μπορούμε δηλαδή να παράσχουμε επαρκή φάρμακα στους Ευρωπαίους πολίτες. Φάρμακα που έχουν δικαίωμα να αποκτούν, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι στις δυτικές χώρες. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω για πιο συγκεκριμένα μέτρα. Στην, ε, στον ανακοινωθέν τύπου σας, σε δήλωση στον τύπο πάντως, μιλήσατε γι' αυτό και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω για την φυματίωση που είναι από τις πιο σοβαρές ασθένειες που μεταδίδεται τώρα στην Ευρώπη και μάλιστα και λόγω των μεταναστευτικών ροών. Ποια είναι τα βήματα που σχεδιάζεται να κάνετε στη διάρκεια της Προεδρίας σας για την καταπολέμηση της χρηματίωσης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον ε, Υπουργό, τον κύριο Τόμας Ντρούκερ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στις ε, φαρμακοβιομηχανίες είναι το θέμα που έχει θίξει και ο Ζιλ Περνιόκ καθώς και άλλοι όσον αφορά τις τιμές των φαρμάκων και την ε, ραγδαία αύξησή τους που εξαντλούν ε, τον προϋπολογισμό μας ε, για τη γιατρική περίθαλψη στα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα ήταν αδύνατο να πετύχουμε διαφάνεια στην τιμολόγηση. Στις Ηνωμένε Πολιτείες έγινε προσπάθεια αλλά με επιτυχία μπλοκαρίστηκαν οι προσπάθειες αυτές για διαφάνεια στην τιμολόγηση. Θα πρέπει στην Ευρώπη να στριμώξουμε τις φαρμακοβιομηχανίες ε, για να γνωρίζουμε ε, ποιες είναι οι δαπάνες τους ε, για τη διάθεση στην αγορά, ποιες είναι οι δαπάνες τους για την έρευνα και ανάπτυξη διότι μεγάλο μέρος της έρευνας χρηματοδοτείται με ε, δημόσιο χρήμα. Χαρίζουμε όμως ε, τις έρευνες αυτές ε, στην βιομηχανία και η βιομηχανία με τη σειρά της αυξάνει τις τιμές. Θα πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το άλλο θέμα είναι επίσης συγκλονιστικό. Έχει καταφέρει η φαρμακοβιομηχανία με δραστηριότητες lobbying να πιέσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ε, ΕΜΑ, ε, ε, στο θέμα των κλινικών δοκιμών. Η φαρμακοβιομηχανία έχει καταφέρει να μπορεί κανείς να διαθέσει στην αγορά φάρμακα με μια γρήγορη διαδικασία όλοι γνωρίζουμε ασθενείς ε, που ε, ε, επιθυμούν διακαώς να λάβουν ένα φάρμακο. Αλλά πρέπει να γίνουν δοκιμές να δούμε βοηθάει το φάρμακο αυτό, σκοτώνει τους ανθρώπους, υπάρχουν παρενέργειες. Η διαδικασία αυτή πιλωτικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έχει συντομεύσει την διαδικασία και έχει γίνει πιο οικονομική. Πιο οικονομική για ποιον στο κάτω-κάτω. Και στην νομοθεσία θεσπίζεται ότι δεν μπορεί κανείς να προσφύγει κατά των φαρμακοβιομηχανιών που ε, διαθέτουν τα προϊόντα στην αγορά. Δηλαδή ακόμα και αυτό το ένα ελεκτικό μέτρο, το ένα αντισταθμιστικό μέτρο που υπάρχει στην Αμερικανική νομοθεσία το έχουμε καταργήσει. Και αυτό είναι εγκληματικό. Είναι σκάνδαλο ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εγκρίνει τη διαδικασία αυτή και θα πρέπει να φροντίσουμε να σταματήσει η διαδικασία αυτή όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι είμαστε έτσι τελείως χαμένοι στην αγορά φαρμάκων. Σας ε, καλώ λοιπόν ε, κύριε Υπουργέ, ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να ασκήσετε πίεση στην Κομισιόν που παραπλανήθηκε. Διότι ναι, οι ασθενείς θέλουν τα φάρμακα, αλλά έχουμε τελικά την κατάσταση να βρισκόμαστε σε μια αγορά όπου δεν γνωρίζουμε καθόλου τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντορνανό. No. She is not here. Όχι, δεν είναι παρούσα. Να παρακαλέσουμε τον Υπουργό να απαντήσει στις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Chcem sa poďakovať za otázky, Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Πολλές από αυτές είναι πολύ σημαντικές. Ας ξεκινήσω από τα θέματα νομοθεσίας. Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και τα in vitro διαγνωστικά βοηθήματα, ε, στις 15 ε, Ιουνίου στον τριμερή διάλογο πετύχαμε συμφωνία ώστε το Σεπτέμβριο μετά την, αφότου θα έχουν μεταφραστεί όλα τα κείμενα σε όλες ε, τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, να μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική συμφωνία. Από τον τριμερή διάλογο προκύπτει υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια ανακοίνωση. Και έτσι θα γνωρίζουμε σε ποια... Μάλλον θα, θα φροντίσω να ενημερωθώ σε τι φάση βρίσκεται η ανακοίνωση αυτή. Όσον αφορά τον κανονισμό 726 και την τροποποίησή του, είναι σημαντικό να αποφύγουμε την επικάλυψη εργασιών. θα πρέπει να φροντίσουμε να καθορίζονται πολύ σαφώς οι αρμοδιότητες. Όσον αφορά τις κατεξουδότηση πράξης, ε, νομίζω θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μέχρι τώρα είχαμε έναν κανονισμό που κάλυπτε δύο τομείς, ενώ τώρα θα έχουμε ξεχωριστή δέσμη μέτρων κτηνιατρικών. όπου θα περιληφθεί ένα μέρος ε, του πεδίου εφαρμογής ε, του κανονισμού 726. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αποφύγουμε να υπάρξει νομικό κενό. Ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής σας με ρώτησε εάν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, μέχρι το τέλος ε, της Προεδρίας μας. Το θέμα αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μας. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με την δέσμη ιατρικών μέτρων. Είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας. Όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα. Το θέμα αυτό έχει πολλές πτυχές. Αφενός υπάρχει η πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και η Ολλανδική Προεδρία έχει κάνει πολλή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό, ιδιαίτερα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Έτσι, η Ολλανδική Προεδρία έχει θέσει τη βάση για τον καθορισμό του προβλήματος. και για την ε, συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά την ε, πολιτική τους απέναντι στις φαρμακοβιομηχανίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα στην ε, βιομηχανία φαρμάκων. οι βιομηχανίες φαρμάκων θέλουν να διαθέσουν στην αγορά πολύ ακρίβα ε, καινοτόμα φάρμακα. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει η σχετική συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου θέλουμε να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή. Θέλουμε να διαπιστώσουμε τι δυνατότητες υπάρχουν όσον αφορά την χρήση αυτών των φαρμάκων. Ξέρετε ότι διάφορα κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένους καταλόγους φαρμάκων ε, και στις χώρες αυτές ε, δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά αυτά τα καινοτόμα φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες στο κάτω-κάτω είναι πολύ σημαντικές για τους ασθενείς. θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνονται επαρκείς κλινικές δοκιμές και τα ευρήματά τους να τεκμηριώνονται επαρκώς. Σημαντικό είναι η ποιότητα ζωής, διότι πολλά φάρμακα απλά παρατείνουν τη ζωή για δύο-τρεις μήνες. Εάν όμως μιλάμε για ε, σημαντική παράταση της ζωής, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, υπάρχει το πρόβλημα των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων. Αυτό είναι πολύπλοκο θέμα, διότι ε, χρειαζόμαστε ελεύθερη διακίνηση των αγαθών. Υπάρχουν όμως χώρες όπου οι τιμές είναι πιο χαμηλές και στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι ασθενείς σε φάρμακα ούτε καν σε γενώσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε λύσεις. και να ξεκινήσουμε συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά. Για παράδειγμα, το κατά πόσο τα φάρμακα είναι εμπορεύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό. Όσον αφορά την οδηγία περί διαφάνειας ε, που ε, ε, απέσυρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, Ήδη από την αρχή τα κράτη-μέλη ήταν κατά της πρότασης αυτής, διότι η οδηγία αυτή αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας και δεν φτάσαμε καν να συζητάμε τις τιμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε την πρόταση αυτή. Όταν όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει νέα πρόταση θα την εξετάσουμε. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ευρύ πεδίο για εθελοντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η τιμολόγηση, η διαμόρφωση των τιμών στον τομέα των φαρμάκων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν ε, υπάρχει πάντα διαφάνεια στο θέμα αυτό, θα πρέπει όμως να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα. όσον αφορά την αδειοδότηση για τα φάρμακα από πλευράς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και τον τρόπο διάθεσης ε, στην αγορά των φαρμάκων. Οι ασθενείς, πολλοί ασθενείς επιθυμούν να έχουν νωρίτερα πρόσβαση σε νέα φάρμακα. Θα πρέπει να εξεταστεί όμως αυτή η συντομευμένη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της Σλοβακής Προεδρίας δεν έχουμε προγραμματίσει συγκεκριμένα μέτρα για το συγκεκριμένο θέμα. Στο παρελθόν υπήρξαν πρωτοβουλίες για την συζήτηση της προσέγγισης αυτής. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται για το θέμα αυτό. Επίσης, στέθηκαν αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή. Μας ρωτήσατε αν θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με την φυματίωση ή αν θα ασχοληθούμε με το θέμα γενικά. Η ενιαία υγεία, η προσέγγιση αυτή είναι σημαντική. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της μικροβιακής αντοχής και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τις αιτίες της μικροβιακής αντοχής ε, στην ε, ανθρώπινη υγεία και την ιατρική. Συχνά συνταγογραφούνται αντιβιωτικά για την ε, καταπολέμηση των ιών. Υπάρχει σημαντικός βαθμός αποτυχίας στην προσέγγιση αυτή. Έτσι υπάρχει λανθασμένη χρήση των φαρμάκων. Εμείς ε, θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στην φυματίωση, διότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τον εμβολιασμό. Επίσης, ε, τέθηκε ερώτηση σχετικά με την ελεύθερη κινητικότητα ε, των ανθρώπων ε, στην Ουκρανία. Το 60% των πασχόντων από φυματίωση πάσχουν από πολυανθεκτικές μορφές της ασθένειας. Θέλουμε λοιπόν ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο για την εφηματίωση ε, για τον ε, ιό του AIDS και για την υπατητή δασέ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής παρόμοιο με το πλαίσιο για την καταπολέμηση του AIDS 2014-2016. Ε, Άλλωστε, πολλοί πάσχοντες από AIDS πάσχουν και από φυματίωση. Βλέπουμε λοιπόν περιπτώσεις Ε, ασθενών ε, με πολυανθεκτικά βακτηριακά στελέχη. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να γίνεται με καλύτερο τρόπο η χορήγηση αντιβιωτικών ε, και στην κτηνοτροφία αλλά και στους ανθρώπους. όσον αφορά την ε, αναγραφή της προέλευσης των κρεάτων στα παρασκευασμένα τρόφιμα. Αυτή η δυνατότητα είναι προαιρετική αυτή τη στιγμή. Έχει εξεταστεί η δυνατότητα υποχρεωτικής αναγραφής. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η λύση αυτή. Τα κράτη-μέλη σήμερα έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν αναγραφή. Η Σλοβακική Προεδρία είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τη συζήτηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δυνατότητα αυτή. Όσον αφορά τη Σύμβαση Πλαίσιο για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού και την σχετική οδηγία. Ε, Ακόμα και αν ε, υπάρξει ε, συμφωνία δεν θα μπορέσει να υπάρξει άμεση εφαρμογή καθότι ε, απαιτούνται ακόμα απαιτείται ακόμα κύρωση της σύμβασης από πολλά κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή μόνο 19 έχουν κυρώσει τη συμφωνία. Στις Βρυξέλλες στις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη, εκδήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο η Επίτροπος Γεωργίευα και ο Επίτροπος Ανδρουκαίτης θα συμμετάσχουν. Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας έχουν οργανώσει τη διάσκεψη αυτή. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκροστέτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Μιλήσατε πολύ για την, τον αγώνα κατά της μικροβιακής αντίστασης και εγώ είμαι η συγκήτρια για τα φάρμακα τα κτηνοτροφικά και χαίρομαι που προσέχετε το θέμα αυτό. Αλλά είπατε ότι θέλετε να προχωρήσετε. Ελπίζω πως μέχρι το τέλος της εντολής θα έχουμε κλείσει το θέμα με το Συμβούλιο, δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε εδώ, γιατί έχουμε χάσει ήδη πολύτιμο χρόνο κατά τη γνώμη μου. Ε, δεύτερο θέμα είναι το θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα. Εσείς προβλέπετε μια μελέτη πλήρη για την ισχύουσα νομοθεσία για τα φάρμακα και για τις προτροπές, δηλαδή τις ευρεσιτεχνίες και τις περιόδους αποκλειστικής ε, άδεια εκμετάλλευσης. Εγώ όμως θα ήθελα να υπάρξουν και μέτρα στήριξης στην καινοτομία, γιατί είναι πολύ σημαντικά και που πραγματικά ε, έχουν αποδείξει την αξία τους μεταξύ άλλων όσον αφορά τα ορφανά φάρμακα φάρμακα. Σας ε, ζητώ λοιπόν να ρημνήσετε ώστε να μην διακινδυνεύσει αυτό γιατί θα διακινδυνεύσει ε, όλη η καινοτομία. Τρίτη παρατήρηση, τα παιδιατρικά φάρμακα όπου θα έχουμε την έκθεση αξιολόγηση της Κομισιόν μετά το καλοκαίρι ε, θέλετε να πιέσετε λίγο ώστε όχι να αναθεωρηθεί ο κανονισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει να γίνουν κάποιες ε, διορθώσεις που είναι απαραίτητε ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί. Ε, τέλος, για την πρόληψη μέσω των εμβολίων, τι μέτρα προβλέπετε για να, να τα κρατημέλη, μάλλον να παροτρύνετε τα κρατημέλη να εμβολιάζουν περισσότερο, κυρίως σε μια χώρα όπως η δική μου η Γαλλία, όπου έχει μείνει πολύ πίσω. Ευχαριστώ. Η κυρία Καμπεθών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και εγώ θα ήθελα να επιμείνω για το θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το κοινοβούλιο μας αυτό. Εσείς αναγνωρίσατε ότι υπάρχει πρόβλημα ανεφοδιασμού, επίσης υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές αλλά και με τις προτεραιότητες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Εγώ θεωρώ, αφού έχω αναλύσει το θέμα, ότι όλα Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει ανεξάρτητα. Πρέπει να υπάρξει μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική για τα φάρμακα. Εσείς αναγνωρίσατε το σημαντικό ρόλο της Ολλανδικής Προεδρίας σε σχέση με αυτό το θέμα και συγκεκριμένα θέλω να τονίσω την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών στις 18 Απριλίου και αυτό που ζητώ είναι να συνεχίσετε και με τη δική σας Προεδρία με το ίδιο ενδιαφέρον όπως και η Ολλανδική Προεδρία ε, να συνεχίσετε την εκθέταση αυτών των θεμάτων. Το Σεπτέμβριο θα υποβάλλουμε ένα σχέδιο που ελπίζουμε πω θα εγκριθεί το Δεκέμβριο με όσο γίνεται μεγαλύτερη πλειοψηφία για το θέμα αυτό. Σα ζητώ λοιπόν να μα βοηθήσετε σε αυτήν την εργασία και συγκεκριμένα να ρωτήσω την ε, σεβασμό ε, μια νομοθεσία που υιοθετήσατε στη χώρα σα το 2014 για το μηχανισμό, δηλαδή θέσπιση των τιμών των φαρμάκων και να βρείτε και έναν τρόπο, να καθιερώσετε έναν τρόπο ώστε να, αναλύσετε, να αναλύετε την θεραπευτική θρησκευτική αξία σε σχέση με τις ζωές που έχουν σωθεί και επίσης σε σύγκριση με τον μέσο μισθό, το μήνυμο μισθό. σα ρωτώ ε, για να ξέρω πώς επηρεάστηκε η προσέγγιση στη, στο θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα από πλευρά των πιο ευάλωτων ομάδων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ριβαζή. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας κύριε Υπουργέ. Είπατε πράγματα σημαντικά. Είπατε ότι σε, σε, μια φάση κλειδί για την Ευρώπη και ξέρετε ότι η υγεία είναι ένα από τα θέματα που οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν ε, η Ευρώπη να ακολουθήσει μια κοινή πολιτική. Υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, είναι στην επικαιρότητα και δεν το αναφέρατε, είναι το πρόβλημα των ενδοκρινικών διατρακτών. Ε, είπατε ότι πρέπει να εξαλειφθούν ή, εν πάση περιπτώσει, να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου. Εδώ ε, έχουμε έναν παράγοντα κινδύνου, τους ενδοκρινικούς διατράκτες, που σύμφωνα με τις μελέτες δείχνουν, όταν μιλήσατε, ας πούμε, για παχυσαρκία, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσει εν μέρη την ε, παχυσαρκία, το διαβήτη, τους διάφορους καρκίνους κτλ. Εγώ θέλω να ξέρω ποια είναι είναι η θέση σας πραγματικά. Είστε με τη μεριά της Επιτροπής, η οποία προσπαθεί να χειραγωγήσει τα κριτήρια και που χειραγώγησε μάλιστα τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να πει ότι είναι μόνο οι άνθρωποι και όχι οι ζωντανοί οργανισμοί. Ή είστε με τη μεριά μας των βουλευτών, γιατί είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς έχετε την Προεδρία αυτή τη στιγμή ε, και ο ρόλος σας θα μπορούσε να είναι καθοριστική σημασία ώστε τα κριτήρια να μπουν στον ορισμό ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλαδή να εξαλειφθούν όλα αυτά τα συστατικά που είναι υπεύθυνα για αυτές τις επιπτώσεις. Ένα άλλο θέμα που δεν προχωρά πολύ η Κομισιόν είναι τα ε, νανοσωματίδια. Ένα σωρό μελέτε έχουν γίνει από ΜΚΟ που δείχνουν υπάρχουν νανοσωματίδιο, διοξίδιο τιτανίου, διοξίδιο πυρητίου, στι τσίχλε, τα μπισκότα και τα λοιπά. Έχουμε μια νομοθεσία που υποχρεώνει στη σήμανση, αλλά και δεν τηρείται. Η Κομισιόν για τα καλλιντικά έπρεπε να κάνει μια έκθεση και ένα, ένα μητρό, ένα αρχείο δεν το έχει κάνει και για τα θέματα που μιλάμε, συζητάμε έχουμε ένα σωρό φάρμακα με μικρο σωματίδια και εμείς δεν έχουμε ιδέα. Και μια τελευταία λέξη για τα φάρμακα και την τιμή αυτών. Δύο τρόποι υπάρχουν. Είτε αυτά που λέτε εσεί, δηλαδή ώστε τα κράτη-μέλη να, ομαδο... να συγκεντρωθούν σε ομάδε και να πιέσουν τι φαρμακοβιομηχανίε και να ορίσουν τα ίδια τι τιμέ των φαρμάκων, ή αλλιώ η υποχρεωτική άδεια. Δηλαδή κάθε χώρα να μπορεί κάλλιστα, η Γαλλία, η στη Τσεχία, η Σλοβακία, να πει εμεί δεν δεχόμαστε την ευρεσιτεχνία, κατασκευάζουμε το συγκεκριμένο αισθητικό από άλλα ε, ε, εργαστήρια, γιατί υπάρχει επίγουσα η ε, ανάγκη για τη δημόσια υγεία και να ορίσουμε έτσι τις τιμές. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντορνανό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ το σχέδιο της Σλοβακικής Προεδρίας φαίνεται να είναι ρεαλιστικό και ισορροπημένο για τα μεγάλα διακυδεύματα της στιγμής από ό,τι άλλες προεδρίες που είχαμε παλιότερα. Όσον αφορά την Επιτροπή μας, θα ήθελα να έχω τη γνώμη σας για τα ζητήματα που μου είναι πολύ ε, προσφυλή. Πρώτον, υγειονομική νομοθεσία που θέλει να προστατεύσει τους εργαζόμενους από τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους ε, φορείς, ε, παράγοντες μάλλον. Ξέρετε την υπόθεση του Αμιάντο που άφησε τα αποτυπώματά της στην κοινωνία. Και έπειτα και, και το και θέμα είναι το θέμα του κινδύνου, του κινδύνου που διατρέχουν ε, οι εργαζόμενοι, οικονομικός και νομικός κίνδυνος για την επιχείρηση και ο κίνδυνος ε, μόλισης για την ε, κοινωνία. Εσείς πού τοποθετείται ε, το κόστος. Το κόστος το οικονομικό ή το κόστος στη δημόσια υγεία. Έπειτα, η σύμβαση πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το καπνό. Πρέπει να στοχεύσουμε τον αγώνα κατά των πλαστών προϊόντων, γιατί υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των φτωχότερων και αυτό λόγω της αύξησης ε, διαρκώς της τιμής του καπνού και προϊόντων καπνού. Ε, συγκεκριμένο παράδειγμα όπου η πολύ έντονη νομοθεσία μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το αυτό που το επιθυμητό. Η Προεδρία σας, κύριε Υπουργέ, θα θίξει αυτό το θέμα και θα αναζητήσει μια ανισορροπία. Τέλος, για θέματα ακόμα πιο καυτά, θα ήθελα να γνωρίζω τη θέση της Προεδρίας σα για τις απειλέ που βαραίνουν το. Ε, αλυσίδα παραγωγής ε, των τροφίμων όπως οι ενδοκρινικοί διατράχτες. Το κείμενο αυτό, το θέμα αυτό μάλλον υπάρχει σε πολλά κείμενα που εργαζόμαστε εδώ επάνω τους και στο μέλλον θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο διαρθωτικό στις ε, πληθυσμούς μας, συσκευασίες, ε, μπογιές και ούτω καθεξής. Είναι μακρύς ο κατάλογος, πρέπει γρήγορα να ληφθούν μέτρα. Τι όθηση θα δώσετε εσείς αυτό το θέμα, ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νικολάσιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Výbor je eh, veľmi, eh, ako vidíte aj z eh. Όπως βλέπετε και από τις ερωτήσεις που σας τέθηκαν, στην ε, Επιτροπή μας υπάρχουν ε, πολλοί ευρωβουλευτές που πραγματικά ε, ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά και τα γνωρίζουν πολύ καλά. Τα θέματα αυτά λοιπόν τα οποία αναφέρατε είναι πολύ σημαντικά για μας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε εδώ και μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξή μας. Τέθηκαν αρκετέ ερωτήσει. Σε κάποιε από εσέ έχετε ήδη απαντήσει. Εγώ θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσει. Η πρώτη είναι η εξή. Η Ολλανδική Προεδρία εστίασε κυρίως στους ασθενείς της νόσου Αλσχάιμερ και γενικά τη γύρανση του πληθυσμού και την γεροντική άνοια. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, διότι είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η Σλοβακική Προεδρία θα θέλαμε να δώσει συνέχεια στις εργασίες αυτές. Μήπως μπορείτε να αναπτύξετε περαιτέρω τα θέματα αυτά. Η δεύτερη μου ερώτηση σχετίζεται με τις μη μεταδοτικές νόσους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας, το οποίο όμως συχνά παραβλέπουμε. Υπάρχουν οι καρδιακές παθήσεις, η παχυσαρκία, η Σλοβακική Προεδρία. Πώς θα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά, ποια είναι η νέα προσέγγιση στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πότ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες ε, από τις ε, ερωτήσεις που ήθελα να θέσω ήδη τέθηκαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σλοβακική Προεδρία ε, για, το, για την πρακτική της αντιμετώπιση. Το περιμέναμε αυτό πολύ καιρό, διότι άλλες προεδρίες ε, δεν ήταν πάντα έτσι. Όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα, διότι θα ήταν καταστροφή να φανταστούμε τη γιατρική περίθαλψη χωρίς χρήση αντιβιωτικών. Αυτό δεν μπορούμε να το φανταστούμε καθόλου. Να σας θυμίσω κάτι που συζητάμε κάθε φορά που μιλάμε για φυτοφάρμακα, τη γλυφοσάτη για παράδειγμα. Φαίνεται ότι κανείς ε, δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι η γλυφοσάτη την οποία χρησιμοποιούμε σε τεράστιες ποσότητες και στην οποία ε, εκθέτουμε ε, μεγάλα μέρη του ευρωπαϊκού πληθυσμού είχε χρησιμοποιηθεί ως αντιβιωτικό. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γλυφοσάτη ήταν ε, για αντιβιωτικό. Ε, η γλυφοσάτη όμως σταμάτησε να χρησιμοποιείται επειδή οδηγεί σε μικροβιακή αντοχή απέναντι και σε άλλα αντιβιωτικά. Εάν ε, λοιπόν εξετάσετε το θέμα της μικροβιακής αντοχής, σας παρακαλώ ε, να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Ε, πολλοί το έχουν παραβλέψει μέχρι τώρα και η Κομισιόν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών και Φαρμάκων παραβλέπουν το θέμα αυτό, αρνούνται να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, δεν έχουν καθόλου ολιστική προσέγγιση. Όσον αφορά τη δεύτερη μερώτηση, είναι και αυτή πολύ σημαντική έχει να κάνει με ε, τις ε, μη μεταδοτικές ασθένειες ε, στις οποίες προτίθεστε να εστιάσετε. Δεν αναφερθήκατε στον διαβήτη. Είναι όμως πολύ σημαντικό αυτό. Σε επίπεδα επιδημίας έχει φτάσει η πάθηση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε επίσης στον τρόπο διαβίωσης και τη διατροφή. Δεν Αναφερθήκατε όμως ε, στην ε, μόλυνση των τροφίμων από φυτοφάρμακα ως αιτία για ε, τα προβλήματα αυτά. Και η κυρία Γκέρλινγκ δυστυχώς αποχώρησε ήδη από την αίθουσα, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ στις δικές της παρατηρήσεις. Συχνά εμείς ως νομοθέτες ελαμβάνουμε αντίθετες ε, γνώμες για το ίδιο θέμα. Έχω μια διαφωνία με την κυρία Γκέρλινγκ στο θέμα αυτό. Της λέω συνέχεια ότι δεν βρισκόμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε ε, ποια επιστημονική γνώμη είναι καλύτερη. Είμαστε εδώ για να αναλάβουμε ευθύνε και να λάβουμε αποφάσεις. Η Προεδρία σας θα πρέπει να ασχοληθεί με το Brexit. Θα πρέπει η Προεδρία σας να ασχοληθεί με τα προβλήματα που βλέπουν οι πολίτες ε, να υπάρχουν. Ε, θα πρέπει να ασχοληθείτε με τις αιτίες του Brexit και σε σχέση με την προηγούμενη μου ερώτηση να αναφερθώ σε ένα μελανό σημείο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τη διαδικασία της επιτροπολογίας και τις εκτελεστικές πράξεις. Σας παρακαλώ να το εξετάσετε αυτό, διότι ε, αν υπάρχει έλλειψη ε, δημοκρατίας, αν υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα σε ένα σημείο της διαδικασίας, τότε αυτό είναι οι εκτελεστικές πράξεις και η διαδικασία της επιτροπολογίας. Εδώ υπάρχει μηδενική δημοκρατία, καμία διαφάνεια και νομίζω θα πρέπει να επιβραδύνουμε ή να ε, ανασχηματίσουμε τη διαδικασία αυτή. Σας παρακαλώ να θίξετε τη συζήτηση αυτή στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Συγγνώμη που μακρηγόρησα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω έναν μετριοπα... μια μετριοπαθή αισιοδοξία γιατί διαβάζω ότι η Σλοβακική Προεδρία θέλει να συνεχίσει την εργασία της Ολλανδικής για την πρόσβαση στα φάρμακα και είδα και από τις προηγούμενες παρεμβάσεις πόσο πολύ μας είναι αυτό το θέμα προσφυλές ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε εκφραστεί και με την ψήφο μας γιατί θεωρούμε πως είναι πραγματικά ουσιαστικό και πρέπει να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα αυτή η υπόθεση της πρόσβασης πρόσβασης, ε, διευκόλυνση στην πρόσβαση, το να έχουμε δηλαδή σύντομες προθεσμίες έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω πώς το λαμβάνει υπόψη αυτή την έντονη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, γιατί έχω την εντύπωση πως αν άκουσα καλά, ότι τα κράτη διστάζουν λίγο, ιδιαίτερα όσον αφορά την μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά αυτό το technology assessment που εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Κάτι ακόμα για το οποίο γενικά ντρεπόμαστε όλοι να μιλάμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που σήμερα τα εφημερίδες, τα μέδια λένε ε, υγειονομική επίγουσα ανάγκη, ε, η ε, συναγερμός, υγειονομικός συναγερμός σε σχέση με τα μετανάστευση. Όμως, αποφεύγοντας να το συζητήσουμε, δεν καθησυχάζουμε τους πολίτες. Υπάρχει όντως πρόβλημα και παγκοσμίω πριν από κάνα δύο χρόνια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε δηλώσει παγκόσμια συναγερμό, υγειονομικό συναγερμό για την πολιομελίτιδα. Και και σε υπάρχει ακόμα στη Συρία, στη Σομαλία, στο Πακιστάν, στην Ιγυρία, χώρες από τις οποίες έρχονται σημαντικές ροές μεταναστών και το συζητήσαμε και πριν και απαντήσατε όσον αφορά τη φυματίωση που και αυτή είναι μια ασθένεια που συσχίζεται με τις συνθήκες τις οποίες ζει ο κόσμος. Εκατομμύρια πρόσφυγες ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ζουν και στις καλύτερες συνθήκες και άρα εκτίθενται περισσότερο σε αυτές τις, ε, τις αρρώστιες. Τα Ηνωμένα Έθνη είχαν κρούσει το κόνοδο του κινδύνου για αυτά τα εκατομμύρια προσφύγων που διατρέχουν πολύ ψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν την φυματίωση και εσείς μιλώσατε και για την, ε, ε, το συνδυασμό AIDS με φυματίωση, κάτι που δυστυχώς συχνά ε, συμβαίνει, γιατί μάλιστα η φυματίωση είναι ο πρώτος, το πρώτο αίτιο θανάτου των θετικών ε, ανθρώπων και στην Αφρική έχει αυξηθεί πολύ η φυματίωση τα τελευταία χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια δεν έγινε τίποτα. Μετά αργήσαμε κάπως να φτιάχνουμε τεστ. Δεν θα, δεν θα ήταν καλό η Ευρώπη να αρχίσει να σκέφτεται από κοινού, να προβληματίζεται από κοινού, να φτιάξει δηλαδή πολιτικές για αυτά τα θέματα που να φτιάχνουν πρωτόκολλα, εν πάση περιπτώσει κοινέ πολιτικές για αυτά τα πράγματα, για το Ελβετικό Κοινοβούλιο έκανε συζήτηση τον περασμένο χρόνο γιατί στο Κιάσο βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι ε, με φυματίωση ξαφνικά. Οπότε χτύπησε ο συναγερμός και το Ελβετικό Κοινοβούλιο συνεδρίασε. Δεν ξέρω μετά τι μέτρα έλαβαν. Ε, Υπήρξε θέμα. Μήπω λοιπόν η Σλοβακική Προεδρία σκέφτεται ότι πρέπει αυτό το θέμα να το εξετάσουμε με αίσθηση ευθύνη και με μεγάλη ακρίβεια, γιατί διαφορετικά θα ε, χτυπάνε οι συναγερμοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα αποσταθεροποιηθεί η αντίληψη που έχει ο κόσμος για το πώς χειρίζεται η Ευρώπη αυτό το τεράστιο πρόβλημα των, μεταναστών, των μεταναστευτικών όρων. Δεν θα θέλαμε να ξεσπάσει κάποια κατάσταση, κάποια αρρώστια. Θα ήταν πραγματικά πολύ, πολύ σοβαρό και πρέπει να το προλάβουμε. Θέλω να ξέρω λοιπόν η Σλοβακική Προεδρία τι γνώμη έχει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η μικροβιακή αντοχή είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Είστε υπέρ της θέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι τα βασικά αντιβιωτικά θα πρέπει να επιφυλάσσονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση. Άλλη ερώτηση για τα τρανς λιπαρά. Αυτά έχουν μεγάλη σημασία, αλλά έχω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Σύμφωνα με υπολογισμούς, 660.000 άνθρωποι πεθαίνουν τον χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από νόσους της στεφανίας, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση τρανς λιπαρών. Ορισμένες επιχειρήσεις έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή ζητώντας το μέγιστο όριο των τρανς λιπαρών στα τρόφιμα να φτάσει τα 2 γραμμάρια στα 100 γραμμάρια τροφής θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να ρυθμιστεί ευρωπαϊκά ή είναι ζήτημα επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Να σας πω την αλήθεια, είμαι αρκετά υπερήφανη για την Ολλανδία. Ακούστηκε συχνά η Ολλανδική Προεδρία σήμερα. Χάρηκα και με τα λόγια του Υπουργού που είπε ότι επιθυμεί να βασιστεί στα πεπραγμένα της Ολλανδικής Προεδρίας. Πολλά από τα θέματα που έχουμε θέσει εμείς εδώ, άλλωστε συζητούνται και από εσά, όπως η μικροβιακή αντοχή και τα φάρμακα. σε νοσοκομεία και οίκους ευγυρία πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Το ίδιο περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν στους ελέγχους... 0,01% των τροφίμων ελέγχονται, ενώ στις κάτω χώρες 0,1%. Πρέπει να υπάρξουν ενιαίες προσεγγίσεις. Τώρα, τα φάρμακα για σπάνιες νόσους. Επίσης σημαντικό θέμα. Επιβάλλονται άλλωστε αυστηρά πρόστιμα όταν φάρμακα οδηγούνται σε σπάνιδα με τεχνητό τρόπο. Αυτά πρέπει να ισχύσουν όμως για όλες τις χώρες μέλη και όχι μόνο για ορισμένες και για το λόγο αυτό χρειάζονται πανευρωπαϊκές προσεγγίσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σα, κύριε Υπουργέ. Πολλά υπόθηκαν ήδη, αλλά θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των ενδοκρινικών διδρακτών. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σε σχέση με την πρόταση που έχει υποβάλει η Κομισιόν για αυτό το θέμα. Θα προχωρήσετε και αυτό πότε. Ε, Πείτε τι πιστεύετε για την προσέγγιση τη Κομισιόν σε σχέση με του ορισμού που έγιναν ε, δεκτοί σε σχέση με τους, τους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού που σημαίνει ε, ε, συνδυασμό με τις ε, κινδύνους, την ακτίμηση κινδύνου ε, όσον αφορά τα βιοκτώνα. συμφωνείτε? Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο. Μεγάλος κατάλογος από ερωτήσεις. Έχετε τώρα την ευκαιρία να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ďakujem Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ερωτήσεις που έχουν πραγματικά επαγγελματικό χαρακτήρα, είναι πολύ αντικειμενικές και μου δείχνουν ότι η υγεία παρόλο που για πολλούς δεν αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα σήμερα, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Οι τομείς για τους οποίους συζητούμε εδώ υπάρχουν όχι μόνο σήμερα, αλλά το ερώτημα, το ζητούμενο είναι πόσο υγιείς θα είναι οι πολίτες στο μέλλον. Θα προσπαθήσω λοιπόν να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις σας και να απαντήσω. Πρώτα για τα τρανς λιπαρά. Θα στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει αξιολόγηση των μέτρων για την διερεύνηση της χρήσης των λιπαρών και κυρίως για τη μείωση της χρήσης αυτής. Μέχρι τέλους του έτους θέλουμε ε, να υπάρχει αξιολόγηση αυτή και η αξιολόγηση αυτή που θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντική για την Σλοβακική Προεδρία. Θα διεξαγάγουμε διάσκεψη άλλωστε για τις μη μεταδοτικές ασθένειες στις 29 του στην Πρατισλάβα. Αναζητώντας συγκεκριμένα συμπεράσματα για την επιρροή που έχουν τα λιπαρά στην ανθρώπινη υγεία. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα όρια για την χρήση των λιπαρών. Πολλές ερωτήσεις σας αναφέρθηκαν στις μη μεταδοτικές ασθένειες. Επ' αυτού έχω να πω το εξή. Θεωρώ το πρόβλημα αυτό ως ένα από τα πιο σημαντικά. διότι έχει άμεση επιρροή στην υγεία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω όχι μόνο σήμερα, αλλά και για τις επόμενες δεκαετίες. Από, αυτές, από αυτά τα συμπεράσματα θα συναγάγουμε και τις λύσεις που πρέπει να δώσουμε. Θα μιλήσουμε και για, τις, ε, για τη γύρανση του πληθυσμού και για τα, τις καρδιακές παθήσεις, τον διαβήτη και άλλες που σχετίζονται με την μεγαλύτερη ηλικία των πολιτών. Αυτά θα χρειαστούν βεβαίω έξτρα κονδύλια. Εάν οι τάσει αυτές συνεχίσουν να διαμορφώνονται όπως σήμερα, θα έχουμε όλο και περισσότερους ασθενείς που θα πάσχουν από τι νόσους αυτές και θα έχουμε λιγότερους ανθρώπους που θα μπορούν να είναι ενεργοί στην αγορά εργασία. Και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικότερε κοινωνικέ επιπτώσει. και θα θίξει βεβαίως και τα δημοσιονομικά των χωρών μελών. Εν προκειμένου πρέπει να υποστηριχθούν τα καινοτόμα φάρμακα, πρέπει να υποστηριχτεί η ιατρική έρευνα, αλλά πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη. Η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν διάφορες ε, γενεσιουργές αιτίε των νόσων αυτών. Μίλησα για την παχυσαρκία, βεβαίως υπάρχουν και άλλες. Για παράδειγμα, η επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, έλλειψη κίνησης, άσκησης στις ζωές των πολιτών, ο τρόπος ζωής και βεβαίως και πρέπει να ασχοληθούμε με την πρωτογενή πρόληψη. Δηλαδή ο κόσμος να αθλείται περισσότερο, να αλλάξει τρόπο ζωής και βεβαίως και διατροφή κάνατε και άλλες ερωτήσεις. Με ρωτήσατε συγκεκριμένα τι θα πρέπει να προτείνουμε στον κόσμο να καταναλώνει ως ε, τρόφιμα. Βέβαια δεν θα συμφωνήσουμε όλοι με τις λύσεις που θα προταθούν, αλλά πιο υγιεινή διατροφή, πιο ποιητική διατροφή, με λιγότερη ζάχαρη, λιγότερο αλάτι, λιγότερα τρανσλιπαρά. Ίσως είναι σωστό να αρχίσει μια συζήτηση για ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να επιβληθούν όρια. Ίσως να μην προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά στη διάρκεια της Προεδρίας μας, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να αρχίσουμε την συζήτηση αυτή, να διερευνήσουμε δηλαδή αν θα είμαστε σε θέση για τα επόμενα 15-20 χρόνια να επιβάλλουμε τα όρια αυτά. Χωρίς να επιβαρυνθούν βέβαια οι παραγωγοί, αλλά από την άλλη μεριά θεσπίζοντας ένα πλαίσιο για να έχουμε υγιεινή διατροφή για τον κόσμο. Έρχομαι σε νόσους όπως άνοια, Alzheimer's. Εκεί προβλέπουμε διάφορες πρωτοβουλίες. Η άνοια θεωρείται προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου θα οργανώσουμε διάσκεψη, γιατί πρόκειται για την επιδημία της τρίτης χιλιετίας. Θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου στην Πρατισλάβα η διάσκεψη αυτή και θα πρέπει να έχει ως στόχο να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Επίσης, να γίνονται έγκαιρα οι διαγνώσεις, να συνεχιστεί η έρευνα για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών. Αυτά σχετικά με ε, το ζήτημα της άνοιας. Σε ό,τι αφορά τα Ολλανδικά συμπεράσματα του Συμβουλίου για την, για την ε, ισορροπία στην αγορά φαρμάκων, οι αποφάσεις της Ολλανδικής Προεδρίας αναφέρονται στο πρόβλημα αυτό με την έννοια ότι είναι σημαντικές βέβαια για όλους μας και χαίρομαι που μπόρεσαν οι χώρες μέλη να καταλήξουν σε συνένεση. Βρήκαμε μια ολοκληρωμένη, καταλήξαμε σε μια ολοκληρωμένη λύση για πολλούς προβληματικούς τομείς για τη συνεργασία σε ό,τι αφορά τον ορισμό των τιμών, τις διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες, και ο προβληματισμός αυτός, και αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη που θα εκφράσω τώρα, ο προβληματισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε αποκλήσεις των συμφερόντων των χωρών μελών, αλλά θα πρέπει σε εθελοντική βάση να αρχίσουμε να προχωρούμε για να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα προς τα εμπρός. Και κάτι που είναι σημαντικό για μας είναι βέβαια τα αποτελέσματα για να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την χορήγηση καινοτόμων φαρμάκων στους ασθενείς. Τέθηκε και το ερώτημα για τα φάρμακα. Έχουμε ένα πρόβλημα για την ώρα για την ταξινόμηση ορισμένων ακριβότερων φαρμάκων για αυτά μιλώ τώρα, αναλύουμε τις δυνατότητες Έχουμε δίκτυ που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει πρώτα να οριστεί. Μιλώ ιδίως για ασθενείς με ογκολογικά προβλήματα, τα συζητούμε αυτά και με τις ενώσεις παραγωγών καινοτόμων φαρμάκων, γιατί θέλουμε καινοτόμες λύσεις για όλες τις χώρες μέλη. για να φτάσουν στις αγορές των χωρών μελών τα καινοτόμα φάρμακα. Μας απασχολεί πολύ το πρόβλημα του καθορισμού των τιμών πρέπει να αναζητήσουμε συνένεση. Εκπροσωπώ βεβαίως την χώρα που ασκεί την Προεδρία, αλλά μιλώ εξ ονόματος όλων των χώρων μελών. Πάντως, η προσωπική μου γνώμη είναι είναι απηχή αυτά που είπα, αλλά βεβαίως οφείλω να μιλώ εξ ονόματος όλων των χώρων μελών. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα για ορφανές νόσους, δεν έχουμε καμιά πληροφορία. Θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση της οδηγίας 141, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό όταν θα έχει κάνει το πρώτο βήμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για τον κανονισμό για τα παιδιατρικά φάρμακα, θα πρέπει να κατατεθεί σχέδιο, να περιλαμβάνει το σχέδιο αυτά, αυτό τα κλινικά συμπεράσματα. Υπάρχει και πίεση βέβαια προς τους παραγωγούς ώστε να κάνουν τεστ των φαρμάκων πραγματικά σε παιδιά. Αλλά όπως είπα, οφείλουμε να αναμένουμε το πρώτο βήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί χωρίς αυτό το Συμβουλίο δεν μπορεί να προχωρήσει. Και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες το θέμα αυτό μου φαίνεται σημαντικό, είναι και ευαίσθητο. Η Κομισιόν στις 15 Ιουνίου κατέθεσε, εξέδωσε μάλλον ανακοίνωση, και τα συμπεράσματα που περιέλαβε σε αυτήν ακόμα δεν έχουν υποβληθεί επισήμως στο Συμβούλιο, ούτε άλλως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα φροντίσουμε να αξιολογηθούν οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εξεταστούν στο επίπεδο του Συμβουλίου και για το ερώτημα για το γλυφοσάτ αυτό είναι κυρίως αρμοδιότητας άλλου συναδελφού μου. Του Υπουργού Περιβάλλοντος δηλαδή. Όμως είναι σημαντικά τα θέματα αυτά βεβαίως για την χρήση ζυζανιοκτώνων και όλα όσα συζητούμε εδώ είναι βεβαίως θέματα που δεν άπτονται μόνο της υγείας, είναι θέματα που θίγουν ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες πλειώνων υπουργών και έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις ταυτόχρονα στην υγεία. Καρκινογόνες ουσίες, προστασία της εργασίας. Για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την προστασία αυτή, η Σλοβακική Προεδρία αυτό το θεωρεί προτεραιότητα να ασχοληθούμε με το πρόβλημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να μειώσει, να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους. Θέλουμε να αυξήσουμε την προστασία των εργαζομένων. Αξιολογώ πολύ θετικά τις προσπάθειες αυτές. Η πρόταση που έχουμε βλάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια περίπλοκη περίοδο διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις των εμπειρογνωμόνων και επ' αυτού πάντως θέλουμε να κάνουμε ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός και να προωθηθεί το θέμα. Στηρίζουμε λοιπόν την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα εμβόλια και τον εμβολιασμό γενικότερα. Ιδίως παιδιών. Και βεβαίως αυτό αφορά και τους παιδιάτρους. Ο εμβολιασμός, ο καταρχήν ενέχει και προβλήματα και αυτό δεν αφορά μονάχα μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε αναπτυχθεί μια ανοσία απέναντι σε ορισμένες νόσους, όπως ε, για τη φυματίωση, Πάντως, σε ό,τι αφορά την, τις προσεγγίσεις των χωρών μελών, υπάρχουν 15 χώρες μέλη όπου ο εμβολιασμό δεν είναι υποχρεωτικός. Θα δραστηριοποιηθούμε λοιπόν και για το πρόβλημα αυτό. διότι η παράληψη του εμβολιασμού μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη θνησιμότητα παιδιών. Γι' αυτό ε, θα εγκύψουμε πολύ σοβαρά στο θέμα αυτό. Βλέπουμε ε, να γίνεται μια εκστρατεία κατά του εμβολιασμού σε διάφορες χώρες μέλη. Πρέπει να αξιολογήσουμε το πρόβλημα πάρα, πάρα πολύ προσεκτικά. Πρέπει να επιστρέψουμε στα εμβόλια, διότι είναι σημαντικό εργαλείο της ιατρικής επιστήμης κατά των μολυσματικών νόσων. Βέβαια από την άλλη μεριά μπορεί να οδηγήσει και σε ανάγκη λήψης λιγότερων φαρμάκων εφόσον το άτομο έχει εμβολιαστεί. Τα αντιβιωτικά συχνά βεβαίως συνταγογραφούνται και σε περιπτώσεις ε, νόσων, ε, ιώσεων δηλαδή, όπου είναι γνωστό ωστόσο ότι τα ε, αντιβιωτικά εκεί δεν προσφέρουν τίποτε. Βεβαίω η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο αγώνα κατά τη ε, μικροβιακή αντοχή. Πρέπει ε, να συνεργαστούν οι διάφοροι τομεί στα πλαίσια του δικτύου One Health Network. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις χώρες μέλη οφείλει να προωθήσει νέο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής αναμένουμε να διεξαχθούν και άλλες συζητήσεις σχετικά στο επίπεδο βέβαια του Συμβουλίου αλλά και στην άτυπη διάσκεψη κορυφής της Μπρατισλάβα. Σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα, στα τρόφιμα, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σχετικά με την επιρροή του στην υγεία. Ε, πρόκειται για προβληματισμό που θα έχει σημαντικές συνέπειες και για το μέλλον. Μέχρι το 2020 θα πρέπει να επανεξετάσουμε, να ξαναγίνει μια αξιολόγηση όλων των ειδικών ή των προσθέτων που φέρουν ε, το ε στην ε, ε, ονοματολογία τους. Ο κύριος Πότσου μου έθεσε μια συγκεκριμένη ερώτηση σε ό,τι αφορά την επιτροπολογία. Έθιξα το θέμα αυτό στα πλαίσια της συζητήσεως του κανονισμού 726 για το πώς θα χειριστούμε το θέμα αυτό. Πρόκειται για θεσμικό πρόβλημα. η συζήτηση που πρέπει να γίνει θα είναι περίπλοκη. Αυτό που είπατε, ότι στη διάρκεια των συζητήσεων εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο θα χρειαστεί να γίνει ένα βήμα προς τη λύση για να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχετίσατε δε αυτό με το Brexit. Αυτά όλα πρέπει να συζητηθούν, όπως είπα άλλωστε στην αρχή. Πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα και να προσεγγίσουμε τους πολίτες προτείνοντας λύσεις που να είναι κατανοητές για τους απλούς ανθρώπους. Χάρη και στη συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή μάλλον εξαιτία των μέσων της μαζικής ενημέρωσης, οφείλω να πω λαμβάνουν οι πολίτες καμιά φορά πληροφορίες που ωστόσο δεν είναι αληθείς. Πάντως, χρειάζεται ευρωπαϊκή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε και Φυσικά θα έχουμε ε, πολύ, πολλά θέματα για συζήτηση στη διάρκεια της παιδείας σας. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας ε, επίσκεψη και ε, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο εξάμεινο. Κλείνουμε τώρα τη συνεδρίασή μας και θα ξαναπούμε στις 3 για την συνέχεια των εργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεργαστούμε αγαστά. Ευχαριστώ. Γεια σας.